Πρόεδρος έχει πρόταση του ΕΛΚ για διορισμό σε επιτροπή. Ο διορισμός θα δημοσιευτεί στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, τότε ο διορισμός θα θεωρηθεί εγκεκριμένος.